κυρία Μινόρδα Κλιβέτη. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτήν την νέα συνάδελφο, η οποία βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορεί να αναλάβει την θέση αυτή. Τα διαπιστευτήριά της δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, αλλά βεβαίως θεωρούμε ότι η κυρία Μιναντόρα Κλειβέτη μπορεί να συνεδριάσει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω για δύο σημαντικά θέματα. Όπως ξέρετε, έγινε μια βίαιη επίθεση τρομοκρατική κατά μιας ε, σχολής, ενός ε, σχολείου στην Ιταλία. Το σχολείο αυτό ονομαζόταν Βοηθιο Φαλκόνε, τον περίφημο δικαστή και βέβαια τα παιδιά που έχασαν τη ζωή του ήταν τα θύματα αυτής της αποτρόπιας επίθεσης. Δύο κορίτσια και πρόκειται για μια επίθεση που ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί η Μελίσσα 16 ετών η οποία πέθανε και η Βερόνικα η οποία βρίσκεται ακόμα μεταξύ ζωής και θανάτου. Πολλά άλλα νεαρά κορίτσια είναι σοβαρά τραυματισμένα. Πρόκειται για θύματα μιας βομβιστικής επίθεσης. Δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ακόμα τις λεπτομέρειες και το πλαίσιο αυτών των επιθέσεων. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε κυρίες και κύριοι είναι ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ, τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη και δύσκολη κατάσταση να αναγκαζόμαστε να ανακοινώσουμε θάνατο δολοφονίες νεαρών παιδιών, νέων. Και πρόκειται για κάτι που βεβαίως εδώ μας ε, οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που παραβιάζεται διαρκώς από αυτούς τους δολοφόνους. Ότι δηλαδή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δολοφονούνται νέα παιδιά, νέοι, αθώα θύματα. Βλέπουμε όμως κυρίες και κύριοι ότι σήμερα διαρκώς αυτή η γραμμή παραβιάζεται και βλέπουμε ότι ο φανατισμός, η βία, θρησκευτικός, ιδεολογικός φανατισμός είτε και απλά εγκληματικές βίες αποτρόπες πράξεις έχουν σαν θύματα παιδιά, νέους και πιστεύω πραγματικά ότι για τέτοιους ανθρώπους, για τέτοιους εγκληματίες δεν μπορούμε να έχουμε καμία επίοικια. Και βεβαίως οι σκέψεις μας σήμερα πηγαίνουν προς όλες αυτές τις οικογένειες των θυμάτων, τους συγγενείς και φίλους Σκεφτόμαστε τη Βερόνικα που δίνει τη μάχη με το θάνατο και όλους τους γονείς, τους καθηγητές, τους δασκάλους, το σχολείο αυτό που σήμερα έχει περάσει αυτήν την τρομερή δοκιμασία. Αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Ιταλία που έχουν πραγματικά τραυματίσει όλη την περιοχή την ίδια ώρα ξέρετε ότι άλλα χώρα και ένας σοβαρός ε, σεισμός. Έχει πληγεί σοβαρά η περιοχή στην περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνα και σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία υπάρχουν 7 τουλάχιστον νεκροί, πολλοί, πολλοί τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να απευθυνθώ στον Ιταλικό λαό, να τους μιλήσω για την αλληλεγγύη μας και στην περιοχή της Εμπίλια Ρωμάνα, αλλά και προς τα θύματα στο Μπρίντιζι. Και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι πρόκειται για ένα λαό που περνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις, ο οποίος είναι συσπηρωμένος. Και πραγματικά στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω την αναγνώριση όλων αυτών των προσπαθεών και να εκφράσουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στον Ιταλικό λαό. Θα σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχω και κάποιες άλλες ανακοινώσεις που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να σας πω ότι έγραψα στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για τα είδη διατροφής και οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας θα δημοσιευθούν στα πρωτόκολλα αυτής της ε, συνεδρίασης. Ο κύριος Χέρμουτ Σόλτ θα αντικαταστήσει τον Μίκαελ Γκούσταυσον με ανακοίνωση